Άλλο ένα σημείο και επίσης σημαντικό. Και το σημείο αυτό ε, λίγο αποσιωπήθηκε έχω την αίσθηση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε ένα στόχο 25% στα πλαστικά μπουκάλια να είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ξέρουμε ότι τα ε, πλαστικά μπουκάλια είναι πρωταθλητής ε, στα σκουπίδια που βρίσκουμε στις ακτές μας και ρηπαίνουν τις ακτές και τους ωκεανούς. Λοιπόν, 25% να είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό και 30% για το 2030. Αυτό είναι καύσιμο για την κυκλική οικονομία. Επίσης, ε, ε, πλαστικά φίλτρα τσιγάρων υπάρχουν και για όσους δεν το γνωρίζουν. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δυστυχώ δεν δέχτηκαν του δικού μα στόχου μείωση, Από την άλλη έχουμε υποχρεωτική σήμανση επιβάλλει στι συσκευασίε των τσιγάρων για προειδοποίηση ε, για το περιβάλλον. Ένα και μόνο από τσίγαρο που πετά στη θάλασσα ε, μπορεί να ρηπάνει από 700 μέχρι 1000 λίτρα νερού. Επίση, συσκευασίε για τα τρόφιμα ε, φιλόδοξη μείωση και βιώσιμη για το 2026. Θελήσαμε αριθμητικά στοιχεία για τους στόχους, δεν το καταφέραμε, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή την ευθύνη τη φέρει ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα στο άρθρο 4 ε, και τα καλό να το πράξουν όπως το κάνουν η Γαλλία, η Βαλονία ή και η Αυστρία ίδια με μια πολύ πρόσφατη και πολύ φιλόδοξη πρόταση του καγκελαρίου Κούρτς. 6,5 δισεκατομμύρια οικονομίες ε, θα έχουμε για τους πολίτες και 30 με 50 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης σε κλάδους που πραγματικά έχουμε τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ περισσότερο από την οδηγία για τα καλαμάκια εντός εισαγωγικών τα σχολαστικά, γιατί έτσι τη βαφτίζουν ε, και την ανάγουν σε αυτό. Ε, επίσης, αναθεώρηση φιλόδοξη προβλέπουμε για τις συσκευασίες με αριθμητικούς στόχους, πρόγραμμα δράσης ευρύτατο απέναντι στα μικροσκοπικά πλαστικά. Τώρα εμείς ασχοληθήκαμε με τα μεγάλα πλαστικά. Και μετά μια ε, πραγματική μετάβαση Ευρώπη Ευρώπης στην κυκλική οικονομία με ε, κλάδους ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. Για τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου ε, να πούμε ότι είναι προϊόν ομαδικής εργασίας αυτό που σας παρουσιάζω. Πρόεδρε, θα πάρω και λίγο χρόνο από τη δευτερολογία μου. Ε, ε, ε, σε ιερή συμμαχία συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ και σας κύριε Τίμερμανς για τη δέσμευσή σας, κύριε Βέλα για τον ενθουσιασμό σας, την Υπουργό Κιόστιγκερ από την Αυστριακή Προεδρία, αλλά και την κυρία Άουκεν, την κυρία Μπόιλαν και τους υπολείπους σκιώδης, Δε Μέσμακερ, Καλ Χάιντς Φλόρενς αλλά κυρίως στους Ευρωπαίους πολίτες, αυτά τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που κινητοποιήθηκαν και μας επίεσαν να βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη για τους ωκεανούς μας φυσικά, για το περιβάλλον, αλλά κυρίως για μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Ρίζ. Και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Τίμερμαν, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απόφαση που θα πάρει σήμερα το Ευρωπαϊκό θα θέσει σε βιώσιμο μονοπάτι την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά. Είναι επίσης απόδειξη ότι ε, ακολουθούμε τις δεσμεύσεις μας. Ποτέ το φυσικό μας περιβάλλον δεν έχει βρεθεί σε τέτοια ε, κατάσταση ε, α, ακραίας έντασης. Η νέα οδηγία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, καταναλώνουμε και κατασκευάζουμε τα πλαστικά. Θα μειώσει την βλάβη προκαλούν στο περιβάλλον πολύ σημαντικά και ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν αλλάζουμε τον τρόπο. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, θα καταστρέψουμε του ωκεανού. Ε, τα επιστημονικά στοιχεία είναι ε, α, α, ε, κατηγορηματικά. Πρέπει να αναλάβουμε εμείς ε, την ηγεσία αυτού του αγώνα αυτής της εκστρατείας. Όπως είπε η κυρία Ρης, πριν από ένα χρόνο όταν ανακοινώσαμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα, για τα πλαστικά, είχαμε πει ότι θα υποβάλουμε αυτή την πρόταση. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει την τελική του απόφαση. Ήδη ε, έχουν δημιουργηθεί πολλές καινούργιες βιώσιμες ε, λύσεις εν ώψη της έγκρισης αυτού του κειμένου, ακόμα και πριν ακόμα εγκριθεί. Ε, μια θετική ψήφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει ένα θετικό μήνυμα στο πλαίσιο της, ε, της στρατηγικής της κυκλικής οικονομίας. Ε, θα γίνουν επενδύσεις σε νέα προϊόντα και θα προωθούν καινούρια επιχειρηματικά μοντέλα. Τα μέτρα αυτά επίσης θα μειώσουν την μόλυνση των υδάτων μας από τα πλαστικά. Θα ήθελα στη Φερντερή Κρίς και στους άλλους κοιόδης ηγητές να απευθυνθώ και να του συγχαρώ. Γιατί και οι τρεις πλευρές ε, του τριμερούς διαλόγου ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν σε ένα θέμα στο οποίο πολλοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε. Συγχαρητήρια, Φρεντερίκ, λοιπόν, και στους υπόλοιπους ε, σκιώδη ηγητέ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου. Ευχαριστώ, Φράνς, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αυτό το νομοθέτημα είναι πολύ αναμενόμενο και πρέπει να στηρίξουμε, ε, να έχει υποστηριχθεί και από πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει όμω να προσβλέψουμε φιλόδοξα μέτρα και να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και στην πράξη. Η πρόληψη τη ε, εξάπλωση των πλαστικών είναι καθήκον των δημόσιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα αξιών και παραγωγή των πλαστικών θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Τα κατάλληλα προϊόντα για το σχεδιασμό των προϊόντων και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών πρέπει τώρα να ληφθούν για να μειωθεί και η κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων εκεί που θα μπορούσαν να υπάρχουν βιωσιμότερε εναλλακτικέ λύσει. Το Ευρωκοινοβούλιο επίση πίεσε να λάβουμε αυστηρά μέτρα για να προβλέψουμε κατάλληλη διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων με επιτάχυνση από την πλευρά των ε, παραγωγών ε, ε, στι διαδικασίε συλλογή και βεβαίω και στον τρόπο κατανάλωση τα μοτίβα κατανάλωση που ακολουθούν οι καταναλωτές, για τα πλαστικά μπουκάλια α πούμε. Εάν περιορίσουμε τη χρήση, του, θα αλλάξει η ίδια η διοργάνωση της οικονομίας. Θα δώσουμε μια όθηση για δευτερογενή ε, υλικά. Επίσης, ε, στηρίζουμε πλήρως τη συμφωνία που επετέφθη στην, ε, στις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να κάνει τρεις δηλώσεις συγκεκριμένα. Ως αρχή ο κανόνα τη μη γνωμοδότηση είναι ότι όταν δεν υπάρχει καμία γνωμοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εξουσιοδότηση πράξη χωρί δικαιολόγηση. Ε, δεύτερο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ε, κατα... εφαρμοστική πράξη από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει να εξετάσει το εφικτό τη στήριξη των προθεσμιών. Και τρίτον, για την περιττή συμπερίληψη ορισμού των βιοδιασπόμενων ε, πλαστικών, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην οδηγία και στην ε, εφαρμογή τη. Ξεκάθαρα θα πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για του κανόνε αυτού, διότι αντιμετωπίζουν τη ρήπανση από τη χρήση των πλαστικών μια χρήση μέχρι και όλε τι άλλε περιπτώσει. Εφόσον εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή, όχι μόνο θα προλάβει την ε, εξάπλωση και την ρήπανση από πλαστικά, αλλά θα γίνουμε και ε, πρωτοπόροι στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότερη πολιτική και στρατηγική για τα πλαστικά. Εδώ το Ευρωκοινοβούλιο ε, διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο για να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για αυτήν την μετάλλαξη στην κοινωνία μα και ελπίζω ότι όλοι θα βοηθήσουμε για να γίνει και πράξη. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Φραν. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια τη Φρεντερίκ Ρη και όλου του σκιώδει εισηγητέ, καθώ και του συνεργάτε μα από τι Γενικέ Διευθύνσει τη Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Και τώρα η κυρία Κάπελ, που δεν βρίσκεται όμω στην αίθουσα. Ο κύριο Ροπέ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, συνάδελφοι, το ζήτημα αυτό είναι ε, ύψης της σημασίας. Έχουμε καθυστερήσει. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους επιτρόπους και την εισηγήτρια αλλά και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου που επέτυχαν μια εξισορροπημένη συμφωνία για να βρεθούν λύσεις. Λύσεις ώστε να περιορίσουμε τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης. Ε, ε ως ε, πρόεδρο, όπως είπε και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης αλλά και των γεωργικών υποθέσεων ε, και στις δύο επιτροπές καθώς και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, υποστηρίχθηκαν οι προτάσεις μου. Δυστυχώς η πρότασή μου αυτή καθεαυτή δεν υπεστηρίχθη μέχρι τέλους για τους συγκεκριμένους στόχους ε, για τα κάτι μελη ως προς την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. Αυτό δεν πέρασε. Υπέρχουν μόνο κάποιες ασαφείς ε, προτάσεις σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπριάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπη, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Τα πλαστικά έχουν αρνητικές συνέπειες για τους φυσικούς μας πόρους και για το φυσικό περιβάλλον. Καταστρέφουν και την αλληλεία και βεβαίως είναι επικίνδυνα και για την ανθρώπινη υγεία. Τα απόβλητα, καθώς διασπώνται, καταλήγουν στην διατροφική αλυσίδα και πολλές φορές και στα τραπέζια μας. Ε, μια πρόσφατη έκθεση του Ocean Cleanup έδειξε ότι η παρουσία πλαστικών στον ελληνικό και δεν είναι μόνη περίπτωση γίνεται το λένε και μεγαλύτερη. Καλύπτει με ε, μια έκταση που είναι τρεις φορές ως η Γαλλία με, χιλιάδε με χιλιάδες ε, τόνους. Θεωρώ ότι εδώ οι αλείς μπορούν να διδαματίσουν σημαντικό ρόλο για την αναχέτηση των πλαστικών και τη εξάπλωσή τη. Και για την ε, αποκομιδή του και για την ε, εξάπλωσή του στη θάλασσα. Το έδειξε και η πρωτοβουλία Fishing for Litter. Ε, και να κλείσω και με την περίπτωση τη Γκρέτα και τα λόγια τη, που λέει ότι χρειαζόμαστε πάντα ελπίδα, αλλά χρειαζόμαστε και δράση. Μόλι ξεκινήσουμε να αναλαμβάνουμε δράση, θα αρχίζουμε να βρίσκουμε και λόγου να ελπίζουμε. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω, γιατί δεν υπάρχει πια χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Λίζε για δύο λεπτά, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η ρήπανση των παγκοσμίων θαλασσών από πλαστικά είναι τεράστιο πρόβλημα, όπως στον Ειρηνικό, που είναι πενταπλάσια η έκταση από την πατρίδα μου τη Γερμανία των πλαστικών στον Ειρηνικό. Χρειάζεται δράση άμεση. Όπου υπάρχει ε, αντίστοιχο υποκατάστατο αντίστοιχης ε, αξίας, ε, έχουμε απαγόρευση. Ε, ας πούμε στα πλαστικά πιάτα. Ε, υπάρχουν χάρτινα πιάτα και ακόμα καλύτερα πιάτα που πλένονται. Και μπορείς να τα χρησιμοποιείς πολλές φορές υπάρχει ε, στρατηγική μείωση σε εκεί που δεν έχουμε ακόμα την απαραίτητη τεχνολογία για υποκατάστατα. Βέβαια, οι στόχοι θα πρέπει να ήταν πιο σαφεί ε, κατά εμέ, τουλάχιστον τώρα να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να του κάνουν όσο γίνεται πιο αυστηρού. Ευχαριστώ όλου εκείνου που βοήθησαν και τη Φρέντερη Ρίξ, ε, αλλά και από το ΕΛΚ τον κύριο Φλόρεν και την ε, Προεδρεύουσα στο Συμβούλιο, την Αυστριακή Υπουργό Ελίζαμπετ Κούστιγκερ, που πραγματικά με μεγάλη δεξιοτεχνία διεύθυνε τι συζητήσει. Χαίρομαι που δεν το παρακάναμε γιατί είχαμε και κάποιες τροπολογίες των ε, πρασίνων που ήθελαν να απαγορεύσουν ε, ε, ακόμα και τα πλαστικά μπαλόνια. εντάξει, να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες και σε καινοτομία, αλλά να μην αφαιρούμε αυτή τη διασκέδαση από τους ανθρώπους. Ε, για τα μικροσκοπικά πλαστικά περιμένουμε νομοθετική πρωτοβουλία για να ασχοληθούμε και με το πρόβλημα αυτό δραστήρια. Σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Ενισχύουμε την κυκλική οικονομία και ε, κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε ε, να γίνουν σκουπιδό οι θάλασσές μας. Σπάνια έχω ζήσει τόσο ανεπιφύλακτα θετική υποδοχή ε, μιας περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον κόσμο. Και πραγματικά μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Θα δεχόσασταν μια μπλε κάρτα από τη συνάδελφό μας την κυρία Μπόιλαν. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λίζε. Είναι χαρούμενος που αυτοί και άλλοι επιτυχημένα ε, ε, απέρριψαν την ιδέα τα πακέτα με τα μπαλόνια να έχουν το, την κατάλληλη σήμανση έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τους ε, καταναλωτές ε, να μην τα απορρίπτουν. Ε, πόσο τρομερό θα ήταν αυτό. Θα συνεχίσουμε τώρα να ζούμε τον τρόμο του περιβάλλοντος γεμάτος μπαλόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να ποντάρουμε στην εναλλακτική τεχνολογία. Ακόμα και η σήμανση και η προειδοποίηση ε, θα σήμαινε ότι να μην χρησιμοποιούμε μπαλόνια σε παιδικά γενέθλια και άλλες γιορτές. Ε, ε, όχι, αυτό το παρακάνει και δεν αφορά καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πρέπει να ποντάρουμε στην καινοτομία και όχι στην απαγόρευση. Και όχι να στείλουμε ε, εδώ ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε τον κόσμο να, να ψυχαγωγείται και να διασκεδάσει. Δύο λεπτά, Παολούτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την θαυμάσια δουλειά της. Ε, αυτή που από κοινού Ολοκληρώσαμε. Συνάδελφοι, νομίζω ότι με την ε, ψήφο μα εντό λίγων ωρών και εγκρίνοντα την οδηγία για την περιορισμό τη χρήση των πλαστικών μια χρήση, θα ε, βοηθήσουμε. Θα βοηθήσουμε να γίνει ένα βήμα προόδου περισσότερη προσοχή στην παραγωγή, περισσότερη διαλογή των απορριμμάτων, περισσότερη ευαισθητοποίηση για του καταναλωτέ και περισσότερε ευθύνε για του παραγωγού. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την ψηφοφορία αυτή που θα μα επιτρέψει δύο σημαντικά βήματα. Πρώτον, να αναχαιτήσουμε την εσφαλμένη νοοτροπία ε, τη αποκομιδή για τον ξέφρενο καταναλωτισμό και την αλόγιστη αποκομιδή και να προστατεύσουμε τι θάλασσε, του βασικότερου πνεύμονε του πλανήτη μα πρέπει να δημιουργήσουμε νοοτροπία κατανάλωση που να βασίζονται στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Βεβαίω δεν εξαρτώνται όλα από την Ευρώπη και μόνο, αλλά η φιλοδοξία τη Ευρώπη μπορεί να γίνει υπόδειγμα. Υπόδειγμα που να δώσει παράδειγμα προ μίμηση σε άλλου, για να γίνουν και άλλα βήματα πρόοδου στη συνέχεια. Άκουσα αυτέ τι ώρε και αυτέ τι μέρε σφαλμένε αντιλήψει ότι η μάχη μα δεν είναι κατά τη ε, βιομηχανία τη χημική που είναι στατικική σημασία για μα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, δεν είμαστε κατά των χημικών. Ε, θέλουμε να γίνουν νέε τεχνολογικέ ανακαλύψει και να αλλάξουν οι συνήθειε των καταναλωτών. Ο μόνο τρόπο για να να δημιουργηθεί και άλλη απασχόληση και να έχουμε και νέες τεχνολογικές λύσεις. Το είπε και η συγκεκριά. Φαινόταν ο στόχος ε, ανέφικτος Κι όμως θα καταφέραμε και μάλιστα σε λίγο χρόνο και με πολύ ευρία στήριξη στο Κοινοβούλιο. Πλειοψηφία και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι και το συμβολικό νόημα αυτής της ψηφοφορία. Έτσι, με αυτό το νομοθέτημα και αυτή την ψηφοφορία θα δώσουμε το μήνυμα ότι η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο επίγουσα αλλά είναι και εφικτή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεμές Μάκερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Την περασμένη Κυριακή για δέκατη φορά έγινε μια μεγάλη δράση καθαρισμού στην φλωμαδική μας ακτή. 7.500 εθελοντές μάζεψαν παρακαλώ 11,5 τόνους, 11,5 τόνους σκουπίδια διπλάσια πλαστικά από ό,τι πέρυσι. Ωραία δράση με συγκεκριμένο αποτέλεσμα που μας φέρνει αντιμέτωπους με το πρόβλημα και το γεγονός. 80% των σκουπιδιών που βρίσκουμε στις ακτές μας ε, είναι πλαστικά και περίπου τα μισά είναι από πλαστικά μιας χρήσεως. Ε, αν δεν υπάρχει ε, ξεδράση, το 2050 θα έχουμε να κολυμπάμε περισσότερα πλαστικά στη θάλασσα από ό,τι ψάρια. Ε, είναι φιλόδοξο λοιπόν αυτό το πακέτο τώρα για να αλλάξουμε ε, ε, την πορεία και να φύγουν τα πλαστικά από τους ωκεανούς. Το πλαστικό είναι πολύτιμο υλικό, αλλά εμείς είμαστε πολύ επιπόλαιοι στη χρήση ε, πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Ε, θα πρέπει ε, να το χρησιμοποιούμε σε όλη την αλυσίδα της αξίας. Αυτό είναι καλό και για το περιβάλλον, και για το κλίμα, και για την οικονομία. Γιατί έτσι αποφεύγουμε εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε τόνος πλαστικού που ανακυκλώνεται ισοδυναμεί σε ένα αυτοκίνητο που θα έφευγε από την κυκλοφορία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πληρώνουν και οι παραγωγή 90% των πλαστικών μπουκαλιών θα πρέπει να συγκεντρώνονται, να συλλέγονται ξεχωριστά. Και επίσης πρέπει να δώσουμε τη μάχη κατά των πλαστικών φίλτρων στα τσιγάρα. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ρής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ωραίο αυτό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ε, ότι αρχίσαμε να τρώμε πλαστικά εδώ και πολύ καιρό. Ο κύριος Τόρβαρτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπή, κυρίες και κύριοι. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα έχουμε πολλές ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και μία από αυτές τις προκλήσεις θα είναι σίγουρα τα πλαστικά. Η συζήτηση αυτή νομίζω ότι ε, μας οδηγεί στην ε, λογική του Σέργιο Λεόνε. Ο καλός, κακός και ο άσχημος δηλαδή. Υπάρχουν καλά πλαστικά αλλά για τους περισσότερους από εμά που χρησιμοποιούμε πλαστικά ε, τα ίδια τα πλαστικά δεν είναι πάντοτε ε, καλά βέβαια. Μερικά χρησιμοποιούνται για να φτιάξουμε γυαλιά οράσεως, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και πλαστικά τα οποία πραγματικά μολύνουν και είναι κακά πλαστικά. Υπάρχουν πολλών ειδών πλαστικά. Αν μπορούσαμε να τα ταξινομήσουμε σε κατηγορίε, ίσως θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι προκλήσει που έχουμε. Για να ξεκινήσει βέβαια κάτι τέτοιο, θα πρέπει να λάβει ε, δράση η Κομισιόν και ελπίζω ότι θα το κάνει στην επόμενη θητεία, ε, κατά τη διάρκεια τη επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Μετά έχουμε βέβαια, όπω είπα και καλά και κακά πλαστικά. Ε, επισκέφθηκα τον Υπουργό περιβάλλοντο τη Νορβηγία που ήταν παλιότερα υπεύθυνο για, για το ε, στάδιο του Όσλο ε, και μου είπε ότι δημιουργούνται τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών ε, όταν κανείς χτίζει ένα γήπεδο. <laughs> Αυτό είναι κακά πλαστικά. Υπάρχουν όμως και καλά πλαστικά. Στην Φιλανδία έχουμε αρχίσει να παράγουμε κύπελα καφέ, για καφέ, χωρίς πλαστικό. Επίσης ε, ε, να παράγουμε πλαστικά διαλυτά, υδατοδιαλυτά, τα οποία πραγματικά μας οδηγούν σε καλύτερη έρευνα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ρίση για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τίμερμαν Δεύτερη, για δεύτερη φορά βλέπουμε ε, νομοθεσία για τη μείωση των πλαστικών. Πρώτα για τις πλαστικές σακούλες, τώρα για ένα μεγάλο αριθμό ε, πλαστικών διαφορετικών τύπων. Είναι σαν να ο αμαρτωλός να είδε ξανά την αλήθεια, να φωτίστηκε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και είναι και πολύ δημοφιλέ θέμα. Έτσι. Δεν είναι παρόλο που δεν σα κατηγορώ για λαϊκισμό. Είναι μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό νομοθετικό κείμενο, αλλά μόνο το πρώτο βήμα. Α το θυμάμαστε αυτό. Είναι κάτι που ελπίζω όμω θα μα οδηγήσει στο να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να δημιουργούμε μόλυνση. Κάθε λεπτό, κάθε λεπτό της μέρας ένα ολόκληρο φορτηγό με πλαστικά χύνεται στους ωκεανούς μας. Βέβαια, ε, η λύση δεν είναι τα βιοπλαστικά ή τα βιοδιασπόμενα πλαστικά, γιατί ακόμα και αυτές οι κατηγορίες πλαστικών είναι φορτωμένες με προβλήματα. Γιατί βιοδιασπόμενα πλαστικά πολύ συχνά ε, διαλύονται σε μικροπλαστικά που και αυτά είναι τρομακτικό πρόβλημα. Ας ε, κερδίσουμε αυτή τη μάχη όλοι μαζί. Ευχαριστώ. το Κύριε Μπόιλαν, θα εγκρίνουμε την ε, οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσεως. Είναι ένα εξαιρετικό νομοθετικό κείμενο. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό χάρη στην εισηγήτρια παρόλο που το Συμβούλιο έχει ε, μειώσει τις ε, ε, αντί όμως ακόμα να αρχίσουμε να γιορτάζουμε, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η βιομηχανία των πλαστικών θα συνεχίσει ε, τη δράση της. Αυτή τη στιγμή απλώς αγγίζουμε την κορυφή του παγόβουνου. Τα μαχαιροπύρων και τα πλαστικά ε, πιάτα είναι μια καλή αρχή, αλλά πού θέλουμε να φτάσουμε, πότε θα σταματήσουμε τα 13 εκατομμύρια τόνους πλαστικών που χύνονται στους ωκεανούς κάθε χρόνο. Ε, η βιομηχανία των ρηκτών καυσίμων και του σχιστολιθικού αερίου είναι αυτή που δημιούργησε αυτή την έκρηξη των πλαστικών. Οπότε αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της, των, της βιομηχανίας των ρηκτών καυσίμων δεν πρόκειται να φτάσουμε και στα πλακτικά. Μιλάμε για την κυκλική οικονομία αλλά θα πρέπει να της δώσουμε σχήμα και μορφή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτή η συνειδητοποίηση για τα πλαστικά μέσω αυτής της οδηγίας, αλλά η απάντηση στην κρίση των πλαστικών δεν είναι η ατομική δράση του κάθε καταναλωτή που ενδεχομένω δεν θα χρησιμοποιεί καλαμάκια, πλαστικά καλαμάκια. Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Ευχαριστώ. Ο Πεντησίνη, ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτέλους, κάποια καλή δύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πολλές φορές ε, την ε, πιέζουν οι πολίτες για να κάνει κάτι που επιθυμούν. Επιτέλους, υποχωρεί στις προσδοκίες των πολιτών. Ε, μια οδηγία θα μας επιτρέψει να έχουμε πιο καθαρές θάλασσες και μέχρι το 2050 να μην έχουμε περισσότερα πλαστικά από ό,τι ψάρια στις θάλασσές μας. Επιτέλους, τα οι συσκευασίε πλαστικών στα σούπερ μάρκετ θα ε, αλλάξουν. Θα υπάρχει εναλλακτική χρήση των πλαστικών, όχι πια τα, τα μια χρήση πλαστικά. Ή τα τσιγάρα από τι παραλίε μα θα πρέπει επιτέλου να πάψουν να εμφανίζονται. Θα πρέπει να επιβληθεί στι ε, καπνοβιομηχανίε να καλύπτουν το κόστο. Το κόστο τη συλλογή, τη μεταφορά και τη επεξεργασία για αυτών των ε, γοπών των ε, υπολοιμάτων τσιγάρων. Θα πρέπει λοιπόν στην οδηγία αυτή να πω ότι δυστυχώ δεν καταφέραμε έναν δεσμευτικό στόχο για να μειώσουμε εντελώς και τα πλαστικά μπουκάλια νερού. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει κάθε χρόνο 50 δις ε, πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά αυτά δεν διασπώνται με το πέρασμα του χρόνου. Σε 20 χρόνια έχουμε 100 δις ε, μπουκάλια να συσσωρεύονται και στις θάλασσές μας. Είναι σκανδαλώδες, διότι οι βουλευτές εμπόδισαν τις καινοτόμες λύσεις των βιοδιασπόμενων πλαστικών, διότι είναι μια καινοτομία που προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την Ιταλία. Νομίζω ότι οι πολιτικέ δυνάμει που υποστήριξαν την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και όσοι την πλόρκαραν, πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του. Ε, δεν επέτρεψε να γίνει ένα ακόμα βήμα ακόμη πιο φιλόδοξο βήμα πρόοδου για ένα καλύτερο περιβάλλον, πιο προστατευμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία, η κυρία Μελά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα ήταν πανίσχυρη και στα χέρια των χημικών. Ε, τους επόμενου δύο αιώνε είχαμε πραγματικέ πρόοδου στην καθημερινή μα ζωή. Δυστυχώ όμω όλα αυτά ε, επλήγησαν από την τεράστια παραγωγικότητα που απέτησε η παγκοσμιοποίηση. Βρισκόμαστε πλέον σε μια ε, κατάσταση δυστυχή, διότι έχουμε τον πλανήτη μα να κατακλείζεται από πλαστικά μια χρήση και στην ξηρά και στη θάλασσα. η, νοικοκυριό ε, γίνεται πάντοτε με πιο γρήγορε ταχύτητε. Υπάρχει βεβαίω κοινωνική εξέλιξη, αλλά είναι προ τον καταναλωτισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να αναλάβουμε δράση για αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα και στι πολιτικέ των κρατών μελών για την έρευνα που θα πρέπει να υποστηριχθεί για να αλλάξουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται και αυτά που διατίθενται στου διανομή και καταναλωτέ, οι οποίοι επίση πρέπει να αναλάβουν περισσότερε αυθύνε και θα πρέπει να παροτρεθούν τα κάτι μέλη να δεσμευτούν. Να δεσμευτούν ότι δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί μια έκτη Ήπειρος που θα αποτελείται από πλαστικά. Ευχαριστούμε η κυρία Γκαρντίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό. Ε, μου φαίνεται σαφές ότι εδώ ε, καταφέραμε να καταργήσουμε τα πλαστικά μια χρήση. Ε, Όπω είπε και ο κ. Πεντητσίνη, λοιπόν, τα άλλα μια χρήση θα επιτρέπονται. Τι θα γίνει λοιπόν με το περιβάλλον μα. Το 25% των πλαστικών που καταλήγουν στου ωκεανού, βάσει μελετών του ΟΗΕ, προέρχονται από εταιρείε τη Αφρική και τη Ασία. Τώρα μην πούμε συγκεκριμένα ονόματα. Όμω είναι ήδη πάρα πολλά. Ε, ένα θέμα που θα έπρεπε να το δούμε με μεγάλη ψυχραιμία, το χρησιμοποιήσαμε ω χαρτί για τι εκλογέ εκλογέ και εσεί, κύριε Τίμερμαν, ω πίτσαν καντιντά των σοσιαλιστών, το χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιείτε και τελικά καταλήγουμε σε κακό αποτέλεσμα. Διότι τώρα δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αυτό ω ε, σημαίακι για να προσελκύσετε Ιταλού. Δεν είναι μετάβαση στην κυκλική οικονομία αυτή. Μιλάτε για απαγόρευση προϊόντων που προέρχονται από την Ιταλία. Και όλε οι άλλε χώρε μα είπαν τι ωραία, μπράβο, δωρεάν όλα αυτά, αλλά τελικά το τίμημα το πληρώνει η Ιταλία τη λύση που επιβάλλεται. Και εγώ δεν πιστεύω ότι τελικά θα πληρώσει μόνο η Ιταλία. Διότι εδώ πραγματικά κοροϊδεύουμε με του ναι. Δηλαδή κάποια καλά στοιχεία τα έχει πρόταση, αλλά όλα αυτά γίνονται όχι με το σωστό τρόπο, ούτε λαμβάνονται υπόψη οι μελέτε τη Πανεπιστημίου τη Καλιφόρνια και του Άλστερ, που λένε ότι τα προϊόντα μια χρήση θα αυξηθούν, θα κυκλοφορούν περισσότερο και θα υπάρχει περισσότερη ρήπανση και στα νοσοκομεία και σε άλλα περιβάλλοντα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ε, σταματήσουμε να εκμεταλλευόμαστε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Ο Γιώργο Λάινεν για μισή λεπτό. 1,5 λεπτό είναι αυτό στα Μα Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά από τη συνάδελφο Γκαρντίνη. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν και κύριε Βέλα, κύριε Επίτροπε, ειλικρινή συγχαρητήρια για την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης. Όπως βλέπετε αυτό που κάνουμε εδώ γνωρίζει μεγάλη αποδοχή ε, το πληθυσμό και είναι και μια ορατή ε, περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά θα πρέπει να το διαφημίζουμε στις ευρωεκλογέ. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, είναι μια ορατή και χειροπιαστή συνεισφορά μας. Προσπαθούμε να ε, καθαρίσουμε το περιβάλλον, να μην γεμίζει σκουπίδια. Ακόμα και αν προέρχονται από άλλες υπήρους σε μεγάλο βαθμό αυτά τα πλαστικά, παρόλα αυτά έχουμε δίκιο που δίνουμε το καλό παράδειγμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν απαγορεύεται και αυτό να είσαι πρωτοπόρος. Και στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική και στη Μεσόγειο καταλήγουν μεγάλα όγκοι ε, αυτού του πλαστικού μιας χρήσης. Η οδηγία αυτή λοιπόν συνεισφέρει και προς τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Ε, να σταματήσει αυτή η κατανάλωση μιας χρήσεως. Χρειαζόμαστε προϊόντα που να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, ε, συχνά ξανά και ξανά, όχι το χρησιμοποιώ και το πετάω. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε πολλά για ε, το σχέδιο, το design των συσκευασιών με πλαστικό, ένα πλαστικό που να μπορεί να ανακυκλώνεται και όχι αυτό το ε, μείγμα τόση μάζα που έχει πρόβλημα στην ανακύκλωση. Έτσι, πραγματικά συνεισφέρουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο στην περιβαλλοντική πολιτική. Ευχαριστώ, ο κύριος Βαντάλεν. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ε, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ πλαστικό καθημερινά γιατί είναι φτηνό ε, για καλό και για κακό και αυξάνονται και τα απόβλητα. Ε, οι ακτές, οι παραλίες, οι θάλασσες, τα ψάρια και τα άλλα θαλάσσια όντα ε, ε, κατακλείζονται. Είναι μια ολόκληρη πλαστική σούπα αυτή που κυκλοφορεί στους ωκεανούς. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να καθαρίσουμε τις ακτές και τις θάλασσές μας. Επίσης, θα πρέπει να μειωθεί και η χρήση αλλά και η παραγωγή πλαστικού. Ξέρετε, το πλαστικό γίνεται από πετρέλαιο. Άρα σήμερα με ένα σπάρο δύο τριγώνια μειώνουμε εκτός από τη μείωση των πλαστικών ε, την εξάρτησή μας από χώρες πετρελοπαραγωγές όπως είναι η Σαλαφιστική Σαουδική Αραβία. Καταπληκτικό αποτέλεσμα και συγχαρητήρια μεγάλα. Ευχαριστώ κύριος Γκερμπράντι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ωραία ε, αυτά ε, που συμφωνούμε και χαιρόμαστε με ομόνια ότι στην Ευρώπη ε, απαγορεύουμε τα πλαστικά μιας χρήσης. Σωστό είναι το αποτέλεσμα, αλλά παραμείνουμε στην αυτοκριτική μας. Τα μέτρα αυτά ήδη είχαν εξαγγελθεί το 2010 σε ένα παγκόσμιο χάρτη για μια Ευρώπη ε, που να χρησιμοποιεί ε, με φιδωλό τρόπο τα πλαστικά. Χρειάστηκε 8 χρόνια αυτό το κείμενο για να βρει την έξοδο του κτηρίου Μπερλεμόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, πραγματικά ε, επίγουσα η κατάσταση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, την πολιτική μας, στην οικονομία, στις μεταφορές, στη συνοχή, στη γεωργία. Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά η νοοτροπία και η τακτική μας. Ωραία λοιπόν αυτή η ομοφωνία και η ομόνια που εκπέμπουμε σήμερα, αλλά θα πρέπει να μεταφέρουμε για να περάσουμε γρηγορότερα σε μια καθαρότερη οικονομία, καθαρή. Ε, κύριε Γκερμπράντι, ο πρόεδρος, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Έθριτζ. Uh, Ευχαριστούμε που δέχεστε την ερώτηση. Η ερώτηση είναι εξή. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αλλαγέ, να βελτιώσουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αλλά η παραγωγή πάντα χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει. Και εσείς το είπατε συνεχώς, ότι, το είπατε πολλές φορές ότι το θέμα βιάζει. Δεν πιστεύετε ότι η πρόταση που έχουμε μπροστά μας θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασία. Και αν ναι, πόσες είναι αποδεκτές. 500, 5.000, 10.000. Πότε θα σταματήσουμε να παίρνουμε μόνο υπόψη τις ανάγκες των κατασκευαστών και των παραγωγών. Ευχαριστώ. Η απάντηση. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα φιλελεύθερο και ένα συντηρητικό. Εγώ πιστεύω σε, μια προ... σε ένα προοδευτικό μέλλον. Αυτή είναι μια ιστορία από το παρελθόν. Πάντοτε μα έλεγαν ότι οι νέε τεχνολογίε θα κοστίσουν θέσει εργασία και τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα μα δημιούργησε ένα πιο λαμπερό μέλλον. Το ίδιο θα κάνει και η καθαρότερη οικονομία. Θα μα δημιουργήσει περισσότερε θέσει εργασία. καλύτερε θέσει εργασία και ω μπόνου και ένα καθαρό πλανήτη. Τι άλλο θέλετε. Ευχαριστούμε. Κύριο Έκχαουτ για ένα λεπτό. Uh, Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Ρίς για την ε, πολύ καλή δουλειά της στην ε, μείωση των πλαστικών μιας χρήσεως. Πολύ καλό θετικό βήμα. Ε, εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε αντιμαχία με την Κομισιόν και το σημαντικό είναι ότι πετυχαίνουμε αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κοιτάξουμε λίγο στο μέλλον. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ο Επίτροπος είπε ότι βρισκόμαστε στο μονοπάτι ενό βιώσιμου μέλλοντος. Ίσως είναι υπερβολική αυτή η ρίση, αυτός ο ισχυρισμό. Πολύ καλά να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το μεγάλο κομμάτι των πλαστικών είναι στις συσκευασίε. Κάποια στιγμή η Κομισιόν πριν από δύο χρόνια αναφέρθηκε ε, ε, στην περίπτωση να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Στην στρατηγική που έχει ανακοινώσει βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν. Συνεπώ, α ε, γιορτάσουμε τη σημερινή στιγμή, αλλά α μα πει και η Κομισιόν ποια είναι και τα επόμενα βήματα που θα κάνει προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή μα από τα πλαστικά. Ευχαριστώ κύριε Σοβαρζέ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μέχρι το 2050 Ακούσαμε ότι θα έχουμε στη θάλασσα περισσότερα πλαστικά από ψάρια. Και το πλαστικό κοντεύει να γίνει η πρώτη απειλή της θαλάσσιας ζωής. Σήμερα 5 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών βρίσκονται στη θάλασσα και στη φύση. Και μέχρι το 2050, αν δεν αλλάξει τίποτα, 30 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών θα παράγονται, που είναι τριπλάσια ποσότητα από όλα τα πλαστικά που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα. Ο πλανήτης μας ουσιαστικά έχει γίνει ο πλανήτης των πλαστικών. Και η καταστροφή αυτή η οικολογική είναι πολύ μεγάλη. Η οδηγία για τα πλαστικά θα μπορούσε να είχε αποτελέσει μία καμπή. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα βηματάκι μόνο προς την καλή κατεύθυνση, ενώ θα χρειαζόταν ε, πλήρης επανάσταση ένα νέο μοντέλο θα έπρεπε να εφεύρουμε χωρίς καθόλου πλαστικά. Κανονικά θα πρέπει να ντρεπόμαστε ε, για την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τον πλανήτη. Και επίσης θα πρέπει να ντρεπόμαστε μπροστά ε, σε αυτά τα είδη ε, που ασφικτιούν από τη δική μας αυτή κουλτούρα όλα πλαστικά και όλα απόβλητα μιας χρήσης. Ο κύριος Έθριτς για δυόμιση λεπτά. Πρόεδρε, νομίζω τα πλαστικά μιας χρήσης και οδηγία τους μεταχειρίζονται αδίκως την συσκευασία ε, για τα τρόφιμα και τα ποτά. Όλα τα άρθρα, τα, μάλλον τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα, τα καλαμάκια, τα φλιτζάνια και ό,τι άλλο παράγεται από πλαστικό, είναι συγκεκριμένα αντικείμενα. Δεν είναι κατηγορία προϊόντων που φτιάχνονται από συγκεκριμένο υλικό. Το EPS είναι το μόνο ε, υλικό που δεν επιτρέπεται στον κατάλογο δεν περιλαμβάνεται μάλλον στον κατάλογο. Όμω οι μελέτε τη Επιτροπή δεν αποδεικνύουν ότι το EPS δεν δημιουργεί προβλήματα στι παραλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σα ίσα. Όλου του είδου τα τρόφιμα και τα ποτά, τα αναψυκτικά που βρίσκονται σε συσκευασίε, ακόμα και EPS, μπορούν να είναι 4 ως 6% των απορριμμάτων που καταλήγουν στις παραλίες. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι η τροπολογία για τα EPS ε, κατέληξε να περάσει μόνο τελευταία στιγμή πριν την ψηφοφορία και δεν συζητήθηκε αρκετά στον επίσημο τριμερή διάλογο. Οι σχετικές πληροφορίες δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν αρκετά για το πολυστερένιο και ε, δεν είναι καθόλου αλήθεια ότι είναι περιορισμένε οι συσκευασίε που χρησιμοποιούν το πολυστερένιο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολλά τα ε, πλαστικά που χρησιμοποιούν μικρά κομμάτια πλαστικού μαζί με το πολυστερένιο. Οπότε ε, και για προϊόντα κατασκευαστικά ε, οικοδομών και για άλλες πλαστικές συσκευασίες το υλικό αυτό είναι επικίνδυνο τα μέτρα μας θα είναι μηδενικής αξίας και οι εταιρείε ε, δεν ε, θα κερδίσουν τίποτα. Ίσα ίσα θα μειωθεί το εισόδημά του και θα χαθούν θέσεις απασχόλησης. Στη δική μου την ε, εκλογική περιφέρεια μέχρι το 2021 θα χάσουμε 250 θέσεις εργασίας εάν αυτή η πρόταση περάσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τουλάχιστον 29 εταιρείε που θα πληγούν απευθεία και είναι χιλιάδε Ευρωπαίοι πολίτε που θα χάσουν το εισόδημά του. Θα πρέπει λοιπόν η απαγόρευση του EPS να, και του Φελιζόλ να ε, λυθούν υπόψη. Εδώ σας έφερα μια σημαία της περιοχής για να καταλάβετε πόσε θέσει δουλειά ε, οι εργασίες θα χαθούν. 200 άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι εξαιτία των δικών σας ε, προτάσεων. Ευχαριστούμε ο κύριος Λαντσίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρήπανση από πλαστικά μιας χρήσης στους ωκεανούς και τις θάλασσες, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε τι μόχλευση ε, θετική μπορεί να έχουμε εδώ. Πρέπει να βρούμε βιώσιμες λύσεις και να επιβάλλουμε την διαφοροποιημένη διαλογή, ε, την επιλεκτική μεροδιαλογή στην Αφρική και την Ασία. Εκείνη είναι υπεύθυνη για τη ρήπανση των θαλασσών. Η Ευρώπη θα συνάπτει ελευθερίες, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες που δεν έχουν καμία πολιτική προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτό συμβαίνει. Λες και δεν βλέπουμε ότι τα γεωγραφικά σύνορα δεν σταματάνε τη ρήπανση στις θάλασσες ε, και στην ξηρά το ίδιο. Ε, παραδόξως, αυτές οι εμπορικές συμφωνίες παροτρύνουν την ε, ενίσχυση της ε, χαμηλού κόστους παραγωγής, χωρίς καμία περιβαλλοντική προστασία και με αθέμητο ανταγωνισμό κατά των επιχειρήσεών μας. Δηλαδή, είμαστε και, και κορόιδα και τελικά χάνουμε. Ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε με άλλο βλέμμα αυτήν την αμφίβολη νομοθεσία που προτείνεται, διότι τις κοντόφθαλμες επιλογές μας θα τις, πληρώνουν, θα τις πληρώσουν καταναλωτές και παραγωγή. Γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε? Ωραία. Παρακαλώ. Συνάδελφε, μας είπατε ένα παραμύθι τώρα. Το έχουμε ακούσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Η Ευρώπη δρά και ενεργεί μόνη της. Όμως, ε, ξέρετε πώς έχει ο παγκόσμιος χάρτης της ανάληψης δράσης. Και είναι χιλιάδε οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που περιμένουν την έγκριση τη νομοθεσία αυτή. Κοιτάξτε, από τι κινήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό που προκύπτει είναι ότι 95% τη ρήπανση τη θάλασσα και του ωκεανού ε, προέρχεται από ε, αφρικανικές αφρικανικέ και ασιατικέ χώρε. Χώρε με τι οποίε συνάπτουμε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών χωρί να ασχολούμαστε καθόλου με την πτυχή τη προστασία του περιβάλλοντο. Ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε με τα δικαιώματα των γυναικών, ούτε με τα εργασιακά δικαιώματα ή την εργασία των ανηλίκων. Εδώ λοιπόν υπάρχει τεράστια αντίφαση ε, στην δράση τη ευρωπαϊκή κοινότητα και αυτό υπογραμμίζω. Δεν μίλησα κατά του περιβάλλοντο. Το πρόβλημα είναι πώ λειτουργεί η τα εργασια των ανηλικων εδω λοιπον υπαρχει τεραστια αντιφαση στην δραση τη ευρωπαικη κοινοτητα και αυτή που είναι δυσλειτουργική. Ευχαριστούμε κυρία Πιετικάινεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα αυτό για το σχεδιασμό τη... και τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα να παραχαιρόμαστε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι βεβαία ότι χρειάζονται και άλλα βήματα για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών. Και μάλιστα θα πέσει η φόρα που έχουμε πάρει ε, όταν αναλάβει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως τα πλαστικά και τα μικρο και νανοπλαστικά είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Ε, και έρχονται και από άλλες πηγές. Χρησιμοποιούνται σε απορριπαντικά, καλλιντικά, στη συσκευασία λιπασμάτων και ούτω καθεξής. Τα τρώμε γιατί είναι μικροσκοπικά στις διαστάσεις τους. Είναι πολλές οι μορφές τους λοιπόν και πρέπει να θυμόμαστε ότι μεγάλο μέρος τους έρχεται και από την ε, βιομηχανία κλωστή Ε, θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δει αυτό και για τις ε, βαφές των υφασμάτων και για τα ελαστικά θα πρέπει να αναλάβει, ναι, να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα πρέπει να συνεχιστεί η σχετική προσπάθεια και στο μέλλον. Ευχαριστούμε η ε, κυρία Νταλή για ένα μισή λεπτό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτριά μας ε, και τους σκιώδεις συγγητές, τον κύριο Παουλούτσι, για παράδειγμα, ε, γιατί συνεργαστήκαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα νομοθετικό κείμενο που θα αντιμετωπίζει ε, το ζήτημα. Κάθε λεπτό ένα φορτηγό με πλαστικά καταλήγει στη θάλασσα, στους ωκεανούς και μέχρι το 2030 το ένα φορτηγό μπορεί να γίνουν δύο. Άρα λοιπόν αυτό το κείμενο είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου, είναι ένα παράδειγμα πολιτικής που αλλάζει τις πρακτικές και την οτροπία. Βοηθάει οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση, ιδιαίτερα οι νέοι και τα παιδιά και βέβαια καταδεικνύει και ποιε είναι οι αναλλακτικέ λύσει. Πιστεύω όμω ότι υπάρχουν τρία θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πλέον. Πρώτον, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών τα οποία θα ανακτούμε από τι θάλασσε. Όπω για παράδειγμα, ε, μια, αυτό το παράδειγμα μια ε, γνωστή μάρκα που παράγει αθλητικά παπούτσια από τα πλαστικά. Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πλαστικά δεν θα φτάνουν καν στη θάλασσα. Ένα σύστημα το οποίο θα ε, ανακυκλώνει τα πλαστικά μπουκάλια νερού σε πλαστικά μπουκάλια νερού είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης ε, θα μπορούσαν τα πλαστικά μπουκάλια, ακόμα και ακόμα καλύτερα, να τα κάνουμε υφάσματα. Τρίτον, θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσει το το πλαστικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εταιρεία που παράγει μαχαιροπύρουνα από άλλε κατηγορίε υλικών, μεταξύ αυτών και υλικά, τα μαχαιροπλήρων τα οποία μπορούν ε, να τα φάνε οι καταναλωτές. Ε, ευχαριστώ. Κάποτε θέλαμε όλοι να φοράμε πλαστικά πουκάμισα στην αρχή της δεκαετίας του 60. Το θυμάμαι αυτό. Ε, κυρία Βιέρινγκ. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρής για το καταπληκτικό αποτέλεσμα Διαπραγματεύθηκα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων από πλευρά των Φιλελευθέρων και με ενδιαφέρει από την αρχή πολύ αυτό το θέμα και το οι απόψεις για το πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα. Είμαι ακράδαντα πεπισμένη και παραμένω ότι το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια τα πλαστικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε εμείς να σταματήσουμε τα πλαστικά μιας χρήσεως, να ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση και τις επαναλημμένες χρήσεις, έτσι ώστε να μειωθεί αυτή η θάλασσα των πλαστικών. Αλλά η πραγματική λύση φυσικά βρίσκεται στην έρευνα και την καινοτομία. Θα πρέπει να βρούμε υλικά ε, που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Ο Ευρωπαίος πολίτης ζητά επιγόντως να βρεθεί δράση και να αναλυφθεί η δράση. Αυτή η οδηγία έρχεται να απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Παρακαλώ του συναδέλφου να το εγκρίνουμε αυτό το κείμενο για να μειωθεί αυτή η σούπα των πλαστικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριβαζή για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχει έρθει η ώρα να τερματίσουμε την εισβολή των πλαστικών μιας χρήσης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια να περιμένουμε. Δεν περνάει η εβδομάδα χωρίς να βλέπουμε ε, μαζικά δελφίνια ή ε, φάλαινες στις ακτές μας νεκρά επειδή είναι η κοιλιά τους γεμάτη πλαστικό μικροπλαστικά, κομφετή πλαστικά κολυμπάνε στη θάλασσα αλλά βρίσκονται και στον αέρα. Ε, δεν θέλουμε πια πολυστηρένιο ε, στι συσκευασίε τροφίμων, φελιζόλ δηλαδή. Τα κράτη-μέλη τώρα δεν έχουν πλέον το ηθικό ε, περιθώριο ε, να αμφιταλαντεύονται. Δεν θα πρέπει να υποκύψουν στις ειρήνες της βιομηχανίας που είναι πάντα έτοιμες να εκβιάσουν την απώλεια θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την οτροπία της μιας χρήσης πετύχαμε τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και του ορυπαίνων πληρώνει. Θα πρέπει να σταματήσει πια αυτή η ασίδωτη κερδοφορία. Κυρία Χάζεμκαμπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και με την κλιματική αλλαγή, η νεολαία μας δείχνει το δρόμο και μας ανακαλεί στην τάξη και για τη σούπα των πλαστικών στους ωκεανούς. Σκεφτείτε λίγο ε, τους νεαρούς ε, ήρωες, τον Μπόγιαν Σλάτ που εφήβρε το Ocean Clean Up ή τη Λίλη 10 ετών με την αποστολή της Plastics Pickup. Παγκοσμίω παίρνει τα ενία πλέον η νεολαία για να σώσει τους ωκεανούς. Μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και με βαθιά ντροπή αυτό, διότι εκείνοι καθαρίζουν τα δικά μας σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία έχουν ρημάξει τους ωκεανούς και τη βιοπικιλότητα. Οι νέοι κανόνες για τα πλαστικά μιας κρίσης είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν είναι φυσικά αρκετό αυτό. Παγκοσμίω βλέπουμε σκουπίδια. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, Mars και Procter Gamble. Αυτές είναι οι μάρκες που βρίσκουμε περισσότερο όταν καθαρίζουν τις ακτές. Πότε θα ασχοληθούμε με αυτούς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, στην κερδοφορία των πολυεθνικών ε, αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιου για ένα λεπτό παρακαλώ. E Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαναγκάζει ε, ε στο Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει προ συγκεκριμένη κατεύθυνση έρευνα. Αν δεχτούμε την οξοβιοδιάσπαση του άρθρου 5, ε, θα ε, παραβούμε τα άρθρα 68-73 του κανονισμού REACH. Ξέρετε την δική σας νομοθεσία, έτσι δεν είναι. Η Κομισιόντρα, σύμφωνα με το άρθρο 69 και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών να εξετάσει τα οξοβιοδιασπόμενα πλαστικά, διότι θεωρεί ότι ενδεχομένω δημιουργούν ε, μικροπλαστικά. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, αλλά τον περασμένο Οκτώβρη ανέφεραν ότι ε, δεν πιστεύουν ότι τέτοιου μικροπλαστικά δημιουργούνται. Αν αυτά χρειαστεί να περιοριστούν. Τα άρθρα 70 και 71 του κανονισμού REACH θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν και να γίνει πρώτα μια δημόσια διαβούλευση ε, και περισσότερες μελέτες. Συνεπώ ε, η αναφορά στα οξοβιοθυσμόνα πλαστικά πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 5 πριν δημοσιευθεί η οδηγία στα, στην επίσημη εφημερίδα, γιατί αλλιώ παραβιάζεται την, τον οργανισμό REACH. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Άουκεν. Μάλιστα. Για να είμαι σύντομη, αρνείστε ότι η οξυδοτική βιοδιάσπαση ε, πολύ μικρά κομμάτια τα πλαστικά. Μετά από 100 χρόνια μπορεί αυτό που λέτε να γίνει. Αλλά η οξοβιοδιάσπαση δεν είναι σαφές ότι δημιουργεί πρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να την απαγορεύσουμε. Αρνείστε ότι η οξοβιοδιάσπαση διασπάπει τα πλαστικά σε μικρότερα πλαστικά. Το αρνούμε. Άλλο η οξοβιοδιάσπαση και άλλο η οξοδιάσπαση. Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε καταστρέφει τα πλαστικά. Δεν είναι πλέον πλαστικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό το είδα και στην πατρίδα μου. Πήρα μια μπλε κάρτα, την έβαλα σε ένα κουτί και μετά από πέντε χρόνια δεν υπήρχε τίποτα εκεί μέσα. Ωραία, τώρα που το λύσαμε αυτό, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελαέ, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, Αγαπητοί συνάδελφοι, η ρήπανση των ωκεανών από τα πλαστικά είναι μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να αναλάβουμε ευθύνε με φιλοδοξία. Νομίζω ότι η συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι καλή. Λαμβάνει υπόψη τι εφικτέ λύσει αντικατάσταση των πλαστικών και μα αναγκάζει να ακολουθήσουμε έναν δρόμο πρόοδου. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ρη, του σκιώδει εισηγητέ για τη δουλειά που έγινε. Δεν θα επαναλάβω τι προτάσει που περιλαμβάνει το κείμενο. Υποστηρίζω το γενικό προσανατολισμό του και πραγματικά εκφράζω την ικανοποίησή μου για την απαγόρευση των οξοδιασπόμενων πλαστικών, διότι η ρήπανση που προκαλούν στην ξηρά και στους ωκεανούς είναι τεράστια. Στο τελικό κείμενο επίσης ευτυχώς προβλέπεται και κάτι άλλο που υποστήριζα τα επόμενα χρόνια το πόσο τα πλαστικά είναι βιοδιασπόμενα σε θαλάσσια περιβάλλοντα να καθοριστεί από την έρευνα και τις επιστημονικές μας πρόοδους. Ευτυχώς γιατί και εταιρείε κατασκευή πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επαναχρησιμοποίηση των βιοδιασπόμενων. Θα πρέπει τα, χρήση τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε να είναι δύο διασπόμενα με καινοτόμε λύσει που θα βρεθούν από εταιρείε και να γίνουν τα πλαστικά δύο πλαστικά, πρώτε ύλε που θα ανακυκλώνονται. Ωστόσο και με όλα τα αυτά μπορούμε και οφείλουμε να τα πάμε και καλύτερα. Ε, αυτό το κείμενο είναι μια αρχή. Είναι καθήκον μα οι φιλοδοξίε μα να συνοδευτούν και από τα απαραίτητα μέσα. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Μποναφέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι νέοι που βγήκαν στους δρόμους όλου του κόσμου τις περασμένες εβδομάδες μας ζήτησαν να αναλάβουμε δράση κατεπηγόντως, να βιαστούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό η Ευρώπη αναλαμβάνει δράση και είναι ένα άλλο σημείο υπέρ του περιβάλλοντο στην καταπολέμηση τη ρήπανση από τα πλαστικά, ιδίω στι θάλασσέ μα. Όχι μόνο στου ωκεανού, αλλά και στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο έχουν δημιουργηθεί τεράστιε νήσοι πλαστικών. Με την οδηγία λοιπόν αυτή απαγορεύουμε τη χρήση των ε, πλαστικών μια χρήση, όπω των πιάτων, των ε, μαχαιροπύρουνων και των καλαμακιών. Ε, και πρέπει στα σούπερ μάρκετ να βρίσκονται συσκευασίε που να είναι ανακυκλούμενε και να μπορούν να, να διατηρηθούν περισσότερο καιρό. Ακόμη και τα πλαστικά που επαναχρησιμοποιούνται στα διάφορα προϊόντα. Θα πρέπει λόγω χάρη να υπάρχει ένα περιεχόμενο για τα αναψυκτικά και τα ποτά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να πούμε ότι γίνεται ένα βήμα με την νομοθεσία αυτή προ την κυκλική οικονομία. Στην Ευρώπη καταλάβαμε πρώτη τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στο θέμα αυτό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο και να ε, βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών μα. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπο καταναλωσή μα, αλλά είναι και ο μόνο δρόμο ε, που έχουμε για το μέλλον. Ευχαριστούμε κύριο Γκαμπού για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ρή ε, και τον κύριο Φλόρεντ που ήταν υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, το κείμενο αυτό αποτελεί πυλώνα τη ε, κυκλική οικονομία μαζί βέβαια με άλλα όπω οι, οι εγκαταστάσει του λιμένε για την υποδοχή. Η κοινή γνώμη είναι πλέον πολύ ευαισθητοποιημένη για το θέμα των αποβλήτων. Μερικοί ζητούν να απαγορευτούν τα πλαστικά αυτά. Ταυτόχρονα όμω, εμεί θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. διότι ε, ακόμα δεν υπάρχουν εναλλακτικέ για όλα. Εμείς ως ομάδα θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τι επενδύσει, προκειμένου η βιομηχανία να καινοτομήσει και να δημιουργήσει εναλλακτικέ πλαστικό να τα αντικαταστήσει με πιο βιώσιμα υλικά. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια μετάβαση προς τέτοιου είδους υλικά τα οποία θα μειώσουν το ίχνος μας, το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον γιατί αυτό το χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Αυτή η μετάβαση προς μια πλήρως κυκλική οικονομία είναι και ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασία με ε, προστιθέμενη αξία ε, και ε, μια ευκαιρία για το μέλλον. Όλοι όσοι θα ψηφίσουν στις 26 Μαΐου θέλουμε να υπερψηφίσουν κόμματα και ομάδες ε, που υποστηρίζουν την έφτακτη μετάβαση προς ε, μια, ε, οικονομή, μια κοινωνία πιο ευαισθητοποιημένη. Ευχαριστώ. Κύριε Χουιβοντολόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε αυτά τα θεωρητικά για τη ρήπανση από τα πλαστικά. Αρκεί να δούμε μια φάλαινα στην Ταϊλάνδη που είχε ε, ε, κατά πιο 85 πλαστικές ε, σακούλες και πέθανε. 250 δισεκατομμύρια μικροπλαστικά έχουμε στον κόσμο. Χαίρομαι λοιπόν που θα απαγορευτούν από το 2021 όλα αυτά τα πλαστικά μιας χρήσης, γιατί αντιπροσωπεύουν το 70% της θαλάσσιας ρήπανσης. παντού ισχωρούν στα ψάρια που τρώμε ακόμα και απειλούν τη βιοπικιλότητα. Είναι το πρώτο βήμα για ένα νέο μοντέλο παραγωγής της κυκλικής οικονομίας. Καλύτερα να καταναλώνουμε και καλύτερα να ανακυκλώνουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Θέλω να επιμείνω στην βιομηχανία των πλαστικών που θα πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο σχέδιο Marshall για τους ωκεανούς. Ο Ριπένων πληρώνει στο κάτω-κάτω. Οι βιομηχανίες εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρούν τη γη μας χωματερή τους. Ε, δεν πρόκειται για την επιβίωση της ε, επόμενης γενιάς ή των επομένων, αλλά της δικιάς μας, γιατί τώρα πρέπει να δράσουμε, αλλιώς θα γίνει μια αναστρέψιμη κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Φιέλνερ, έχει το λόγο. Η μείωση των ε, πλαστικών ιδιαίτερα στους ωκεανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό το 85% των αποβλήτων που βρίσκουμε στους ωκεανούς είναι πλαστικά. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές ως προς τις προσδοκίες μας. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση που εγκρίνουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά τα νησιά από πλαστικά μέσα στους ωκεανούς, ε, ούτε και, να, και παραλίες οι οποίες ε, δεν θα ε, υπόκεινται, δεν θα υφίστανται επιθέσεις από κύματα πλαστικών. Τα περισσότερα πλαστικά που καταλήγουν στους ωκεανούς προέρχονται από την Ασία. Πέντε χώρες της ε, Ασίας αντιπροσωπεύουν το 60% τη μόλυνσης από πλαστικά στι θάλασσε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευθύνη. Το αντίθετο, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να δείξουμε το δρόμο στους υπόλοιπου. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κάνουμε εμεί τόσο σωστό πρώτα. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε τι ε, κατάλληλε πηγέ πλαστικών. Ε,